Pan Ας ξεκινήσουμε με μία σύντομη ανακοίνωση. Καταδικάζω την επίθεση της δημοκρατικής, δημοκρατίας της Κορέας εναντίον του νοτίου νησιού Young Πιέντ και καταδικάζω τα σημερινά γεγονότα στην Κορεατική Χερσόνης διότι η χρήση της βίας δεν λύνει κανένα πρόβλημα και ε, πρέπει να αποφευθούν περαιτέρω απώλειες ζωής. Προς όφελος της Κορεατικής Χερσονήσου θα πρέπει ο Βορράς και ο Νότος να προσπαθήσουν να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη σε μια πιο μόνιμη βάση και γι' αυτό και ε, ελπίζω ότι θα αποφευθεί μια κλιμάκωση της κατάστασης. Απευθύνομαι στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας κατά τρόπον ώστε άμεσα να σταματήσει όλες τις εχθρικές ενέργειες και να αποφύγει ε, κάθε ε, κίνηση η οποία θα οδηγήσει σε κλιμάκωση. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή η συμφωνία από την ε, Δημοκρατία της Βορείου Κορέας. Λαϊκή Δημοκρατία της Βορείου Κορέας. Και τώρα